Καλημέρα. Καλημέρα. Επιτρέψτε μου να σας ζητήσω πρώτα απ' όλα να καθίσετε στις θέσεις σας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Με μεγάλη χαρά σας δίνουμε την δυνατότητα εδώ να τα λέτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να χαιρετήσω εδώ όλους τους παρόντες. Την συμπρόεδρό μου πρώτα απ' όλα, εδώ στην έδρα, την ε, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, της χώρας δηλαδή που έχει την Προεδρία. Θα τροποποιηθεί ελαφρά το πρόγραμμά μας. Ο κύριος Ορλάντο Τετοροβίτσι δεν θα είναι εδώ, που είναι ο πρόεδρος οικονομικών και πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, ο κύριος Τεοντρότσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σύγκληση, την σταθερότητα και την συνοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και ποιος είναι ο ρόλος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας γιατί μας επιτρέπει έτσι να προχωρήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δουλέψει και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της θητείας του και ήδη στην Ολομέλεια του Ενωρίου θέτησε τη θέση του για ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα στηρίξει τις επενδύσεις και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το 2021 μέχρι και το 2027. Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να βελτιώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε τα κενά και με τον τρόπο αυτό να πετύχουμε καλύτερες συμφωνίες και να πετύχουμε περισσότερο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Οι Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμών άρχισαν να δουλεύουν πάνω στην πρόταση για θερθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πάνω στη λειτουργία σταθεροποίησης των χρηματοδοτήσεων. Και τα αποτελέσματα τα περιμένουμε τον Μάρτιο. Οι προτάσει αυτές θα αποτελέσουν και την ευριακή μορφή του προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Τέλος, το Συμβούλιο προχωράει πάρα πολύ αργά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη ετοιμάζει μια προσωρινή έκθεση για να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα δώσει συνέχεια στον μηχανισμό σταθερότητας. Και το Κοινοβούλιο δίνει σήματα έτσι στο, στο Συμβούλιο και του ζητάει να προχωρήσει πιο γρήγορα στην εμβάθυνση της ΟΝΕ. Οι προθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να γίνουν κατανοητές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να στηριχθούν. Οπότε, περιμένουμε από εσά να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις σχετικά και να μπορέσουμε έτσι να συνεργαστούμε. Η συζήτησή μας Βέβαια πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, έχουμε ήδη κάποια καθυστέρηση. Και αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε και εμείς να σας κατευθύνουμε για να μην καθυστερήσουμε περισσότερο. Θα σας πω πώς θα προχωρήσουν, πώς μπορείτε να παίρνετε το λόγο πρώτα απ' όλα. Υπογραμμίζω ότι ως ήθιστε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι όσο γίνεται περισσότεροι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ακόμα και αν έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Και ακριβώς επειδή είναι πολλοί συμμετέχοντες, παρακαλώ να καταλάβετε ότι μετά από τις αγωγικές παρατηρήσεις, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι δυνατόν να μπορέσετε όλοι να πάρετε το λόγο σήμερα. Και γι' αυτό ε, σας ζητούμε, όσοι πάρετε το λόγο, να είσαστε σύντομοι, να περιοριστείτε σε 2-3 λεπτά το πολύ. Είναι ο συνήθις κανόνας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Σώμα. Εμείς μερικές φορές δεν έχουμε πάνω από ένα λεπτό και σίγουρα όχι πάνω από τέσσερα λεπτά. Οπότε προσπαθήστε κι εσείς να προσαρμοστείτε. Τώρα, ανάλογα με το πώ θα εξελιχθούν οι συζητήσει, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε το χρόνο και να τον περιορίσουμε ακόμα περισσότερο. Ε, μπροστά σα θα έχετε τις ε, κάρτε που πρέπει να συμπληρώσετε, κάποια μικρά έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε για να καταλάβουμε ότι θέλετε να πάρετε το λόγο συμπληρώστε τις καρτέλες αυτές, κάντε νόημα στους ε, κλητήρες, όποιο κλητήρα βλέπετε στην αίθουσα και εκείνο θα μας φέρει τις κάρτες εδώ στο Προεδρείο. Προσπαθούμε να μοιράσουμε και το χρόνο ομιλία ω εξή. Δύο εθνικοί, ευρω... εθνικοί βουλευτές πρώτα και μετά ένας ευρωβουλευτές. Πάλι δύο εθνικοί βουλευτές, ένα ευρωβουλευτή και ούτω καθεξής. Και όπω είπαμε, ανάλογα χρειαστεί θα προσαρμόσουμε τους χρόνους. Οπότε, κυρία Κάρμεν Λένα Μιχαλτσέσκου, σας καλωσορίζω και πάλι. Είναι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της ε, Ρουμανίας και θα συντονίσει το πρώτο νόημα της συζήτησης. Οπότε, έχετε το λόγο και θα αναλάβετε το συντονισμό, έτσι. Θα φροντίσετε για τους χρόνους κλπ. Και πολύ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας και τον κύριο Έτιγκερ εδώ, που είναι ε, από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, ομιλητές. Η Ρουμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμβάθυνση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, γνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα και όλα τα μέτρα που προωθούν το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η Ρουμανία πάντα έλεγε ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωζώνη, να διασφαλιστεί η σταθερότητα ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας και ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν τονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει τους στόχους αυτής είναι κάτι που δεν πρέπει να διχάζει τις χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη και αυτές που είναι εκτός. Κατανοούμε βέβαια τις ειδικέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρωζώνης, αλλά συγχρόνως υπογραμμίζουμε ότι η σύγκληση είναι κάτι αναγκαίο για όλες τις χώρες μέλη, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Brexit. Η ενότητα είναι θεμελιώδες στοιχείο. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να συμμετέχουν στη διαδικασία όλες οι χώρες μέλη. Οι ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις απαιτούν μεταρρυθμίσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απαιτούν προσπάθεια από όλου. Υπάρχει αλληλεξάρτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποφάσεις για την παγίωση της ΟΝΕ είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε ένα ευρύ σχέδιο που να τους περιλαμβάνει όλους. Αυτό ήταν ε, το σύντομο μήνυμά μου. Με πολύ χαρά λοιπόν συμπροεδρεύω και εγώ την ε, συνεδρίαση αυτή. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ε, παρουσιάσω τον πρώτο εξέχοντα ομιλητή μας, που είναι ο κύριος Γκούντερ Έτιγκερ, Επίτροπος Αρμόδιος για τον Προπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους. Κύριε Έτιγκερ, έχετε τον λόγο. Ξέρετε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την εξέλιξη δύο μεγάλων εγχειρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, το δημοσιονομικό μας πλαίσιο για το 2021 με 2027. Δεύτερον, το εγχείρημα της εμβάθυνσης και της εδραίωσης της Ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Νομίσματος. Και τα δύο αυτά είναι συνειφασμένα στενά μεταξύ τους. Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για το δημοσιονομικό πλαίσιο με τις προδιαγραφές για την επεξεργασία των θεμάτων, τις 37 προτάσεις δηλαδή, για την επεξεργασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τις κατευθύνσεις που στη συνέχεια ανέλαβαν να διαπραγματευτούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Πλευράς του. Η Νομισματική Ένωση λοιπόν έχει να κάνει με μια σαφή δήλωση αναγνώριση τη σημασία του ευρώ. Εάν δούμε πόση δύναμη έχει στην παγκόσμια αγορά το ευρώ, εάν δούμε πόσο μπορεί ο Τραμπ χάρη στο δολάριο να κάνει ε, διεθνή πολιτική, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ζητάει να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα. Έχουμε λοιπόν στο ευρώ, ασχέτως κάποιων προσπαθειών που μπορεί να έχουν επιχειρήσει να το αποδυναμώσουν, το δεύτερο σε δύναμη κράτος. 19 είναι τα κράτη που ανήκουν πλέον στην Ευρωζώνη. Η δύναμή του είναι πολύ μεγάλη. Από το 8, το 9, το 10 και το 11 ε, διαπιστώσαμε ότι το ευρώ έχει αδυναμίες και έκτοτε έχουν αληφθεί πολλές προσπάθειες, παρότι θα χρειαστούν πολλές ακόμη και στα επόμενα, στους επόμενους μήνες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε την, ε, το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής πολύ πιο στενό από ό,τι πριν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που παρακολουθούν τα κράτη-μέλη ε, χρόνο με το χρόνο την με την τήρηση των ε, ιδιαίτερων ανακράτως συνθήκων και προδιαγραφών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, με την Τραπεζική Ένωση η οποία έχει μπορέσει να περιορίσει σημαντικά τους κινδύνους για τον τραπεζικό τομέα γενικά, πολύ περισσότερο από στο παρελθόν, με τον μηχανισμό σταθεροποίησης που αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει σε κατάσταση ανάγκης όπως συνέβη με την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Κύπρο σε ένα βαθμό με την Ισπανία γιατί ήταν απαραίτητο αυτό και επίσης για την ε, Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την ε, Κύπρο χωρίς ε, περιορισμούς στους εθνικούς προϋπολογισμούς, χωρίς δυσκολίες ή συνέπειες στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η Ελλάδα επίσης κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες, αλλά πρέπει να πούμε ότι όταν έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, ένα μόνο νόμισμα σε εποχές ε, εθνικής... Ε, ε, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν έχει κανείς το εθνικό του νόμισμα μπορεί σε περίοδο προβλημάτων οικονομικών να το υποτιμήσει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει βέβαια όταν είναι μέλος της Ευρωζώνης και γι' αυτό υπάρχει η πρόταση για την ανάπτυξη κάποιων ιδιαίτερων εργαλείων για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Και έτσι λοιπόν επιτρέψτε μου για να αναπτύξω αυτή την ε, θεματολογία και τα επιχειρήματά μου να γυρίσω λίγο πίσω στην ιστορία γιατί έχουμε τρεις ομάδες κρατών μελών στην Ευρωζώνη. Η μία ομάδα η οποία επιδιώκει την ε, ε, διατύπωση ειδικού προϋπολογισμού, κατάρτιση ειδικού προπολογισμού για την Ευρωζώνη με τη Γαλλία πρώτη, ορισμένα κράτη της Νότιας Ευρώπης, τη Γερμανία που σε ένα βαθμό ακολουθεί τις προτάσεις του Πρόεδρου Μακρόν. Μια δεύτερη ομάδα η οποία έχει ε, αμυντική και να μην πω αρνητική στάση είναι η ομάδα των ε, κρατών του Βίζιγκρατη της Χάνζα και λοιπόν μια τρίτη ομάδα με κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της ε, Ευρωζώνης και που ως εκ τούτου φοβούνται ότι τα 19 κράτη της Ευρωζώνης θα απορροφούν κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή αυτά τα οποία θα χρειαστούν ενδεχομένως τα 27-28 κράτη-μέλη στα επόμενα χρόνια για την διαρθρωτική πολιτική, τη ιωρική πολιτική, τις υποδομές κτλ η, το Euro Summit, δηλαδή η Σύνοδος Κορυφής ε, των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των Κρατών της Ευρωζώνης, ε, το αποφάσισα πριν από μερικού μήνες, να διατυπωθεί μια συγκεκριμένη στοχευμένη πρόταση για συγκεκριμένα εργαλεία για τα κράτη της Ευρωζώνης, που όμως θα εγγράφεται μέσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό των 27. Και αυτή είναι και η δουλειά που γίνεται τώρα στην Ευρωζώνη από κοινού με τον Υπουργό των Οικονομικών της Πορτογαλίας που είναι πρόεδρος της ομάδας της Ευρωζώνης. Και έτσι, τον Ιούνιο του 2019, η προσεχή Σύνοδος Κορυφή τη Ευρωζώνης μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δουν την κατάθεση των προτάσεων αυτών ο συνάδελφο Δομπρόφσκη ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο ε, Μοσκοβισή επίσης και ο υποφαινόμενο, έχουμε συνεργαστεί ενεργά στην ε, κατεύθυνση αυτή. Δύο εργαλεία λοιπόν έχουμε να προτείνουμε. Καταρχάς, ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα, πρόγραμμα δηλαδή για τον προπολογισμό που θα στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με εργαλεία ε, υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων τα οποία, τις οποίες τα κράτη-μέλη προς το δικό του συμφέρον αλλά και προς το συνολικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εισαγάγουν για να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις με απελευθέρωση της αγοράς, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γιατί ακόμα και έτσι ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, δημοσιονομική υποστήριξη με το εργαλείο αυτό υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Χάρη στο εργαλείο αυτό. Και επίσης ε, θα έχει και μια λειτουργία σταθεροποίηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά κίνδυνο ε, περιστασιακών κλειδονισμών, εάν ε, παραδείγματι ένα κράτος ε, εμφανίσει υπερβολικό κρατικό χρέος. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε να γίνει ένα Brexit χωρί συμφωνία, το τη μεγαλύτερη ζημιά θα την υποστεί η Ιρλανδία μεταξύ των 27 κρατών μελών. Γιατί η οικονομία της Ιρλανδίας είναι πολύ στενά συνδεδεμένη, πολύ στενότερα από οποιαδήποτε άλλη εθνική οικονομία με την Βόρεια Ιρλανδία, καταρχάς και ως εκ τούτου με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν θα κινδύνευε σε μια τέτοια περίπτωση από ύφεση, από ένα κλειδονισμό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε, αν υπάρχει αυτό το εργαλείο, να προσφερθεί δημοσιονομική βοήθεια και να στηριχθούν οι επενδύσεις μέσα από αυτό το ε, εργαλείο σταθεροποίησης με συγχρηματοδότηση. Ένα άλλο παράδειγμα. Για τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλουμε να αποσυνδέσουμε τα συστήματα, τα, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των πιο βαλτικών κρατών από αυτό της Ρωσίας, κατά τρόπο σταδιακό βεβαίως, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίπεινα κυρώσεις Και, τα λοιπά. και τότε τα τρία αυτά όμορφα κράτη, Λετωνία, Λιθουανία και Εσθονία, θα κινδυνεύαν από τι πιέσει τη ρωσική οικονομία. Και αυτό πάλι θα ήταν ένα κλειδονισμό. και άρα θα χρειαζόταν μια ε, προσπάθεια ε, σταθεροποίηση με επενδύσει που θα συγχρηματοδοτούνταν από αυτό το ευρωπαϊκό μέσο. Έτσι λοιπόν δεν θέλουμε έναν ξεχωριστό προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Αλλά αυτά τα δύο εργαλεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, θα μπορούσαν να προσφέρουν καταρχάς εξασφάλιση στην ενότητα του νομίσματος και να δραστηριοποιούνταν μέσα στην Ευρωζώνη κατά τρόπο ώστε να μπορούν τα 19 κράτη της Ευρωζώνης να τα αξιοποιούν, αλλά ταυτόχρονα και τα κράτη τα οποία δεν είναι ακόμα μέλη, αλλά έχουν πάρει το δρόμο της Ευρωζώνης, συγκεκριμένα η Βουλγαρία ή η Κροατία, να, ε, η Ρουμανία επίσης, να μπορούν να στηριχθούν χάρη σε αυτά τα μέσα. Τις προτάσεις αυτές λοιπόν εμείς σκοπεύουμε να τις καταθέσουμε τον Ιούνιο στην Ευρωζώνη, στην Ευρωομάδα, αφού τις ε, ε, συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συλλογικό όργανο έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση λόγω της εισαγωγής αυτών των εργαλείων στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα πρέπει να εγκριθεί φέτος το φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν και θεωρώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή. Παρά τα δύο αυτά εργαλεία ο κύριο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα με τα κύρια εργαλεία του που είναι η πολιτική συνοχή, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι το Μέσον Συνδέοντα την Ευρώπη, που είναι ε, ορίζον 2020 και ούτω καθεξής. Ορίζον Ευρώπη μάλλον. Και εδώ χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη γιατί το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώπης απαιτεί και ομοφωνία. Χρειάζομαι δηλαδή και τους 27 υπουργούς των οικονομικών και τους 27 υπουργούς ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και χρειάζομαι την υποστήριξη και των 27 εθνικών κοινοβουλίων, τη δική σας δηλαδή υποστήριξη. Και γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω να αναλάβετε ενεργό ρόλο και δράση στα εθνικά σας κοινοβούλια, ε, να παρακολουθήσετε τα θέματα αυτά και το τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω. Τον Ιούνιο του 2011 είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις προτάσεις της για την περίοδο μέχρι το 2020, αλλά το Συμβούλιο δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία, δεν αποφάσισε τίποτα. Η απόφαση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ήρθε μόλις το Δεκέμβριο του 2013 και ήταν πια πολύ αργά. Και γιατί, διότι στο χώρο της συνοχής, στο δεύτερο πυλώνα της γεωργίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της ανάπτυξης πέθρου, χρειαζόμαστε συμφωνίε εταιρική σχέση. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί ο προπολογισμό και μόνο τότε μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τι κυβερνήσει ε, των κρατών μελών σε ένα βαθμό, μάλιστα και με τι περιφερειακέ κυβερνήσει, τοπικέ κυβερνήσει, ε, για να συζητήσει και να συμφωνήσει ε, έργα συγκεκριμένα και προγράμματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους γιατί άλλες ανάγκες έχει η Κύπρος, άλλες η Ιρλανδία, άλλες η Πορτογαλία, άλλες η Εσθονία, άλλες η, η Γερμανία, άλλες η Ρουμανία. Και άρα λοιπόν αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέση για να κλείσουν χρειάζονται και ένα χρόνο συνομιλίε. Έτσι λοιπόν το 2015, το 2016 χρειάστηκε να χαρακτηριστούν ω τελείω χαμένο χρόνο εν τέλει, διότι δεν αξιοποιήθηκαν για τα προγράμματα αυτά τη περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν το 20, το 21 και μάλιστα σε μια περίοδο δύσκολη, δεινή οικονομικά, με κράτη που ήδη έχουν μπει όχι μόνο σε στασιμότητα αλλά και σε ύφεση ακόμη, δεν μπορούν να πάνε χαμένα αυτά τα δύο χρόνια, το 20 και το 21. Πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία, πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Το αργότερο λοιπόν μέσα στο τέλος του 2019 πρέπει αυτά όλα να κλείσουν και γι' αυτό το φθινόπωρο του 2019 ανέφερα νωρίτερα ως ημερομηνία. Το 2000, Ιούνιο του 2019 γίνονται οι προτάσεις, το ε, φθινόπωρο κλείνει Πρέπει να κλείσει δηλαδή το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη πέντα αιτία. και σας καλώ εσάς ως βουλευτές των εθνικών σας ε, επιτροπών προϋπολογισμού από τα εθνικά σας κοινοβούλια να συμβάλλετε κι εσείς εγκαίρως να κλείσει αυτή η δουλειά, να προσφέρετε την, ε, τη δουλειά και την υποστήριξη σας βεβαίως. Σήμερα έχουμε το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων που συνεδριάσει υπό την ε, Ρουμανική Προεδρία. Σε μερικά λεπτά, σε μερικά δεκάλεπτα πρέπει να πάω εκεί για να παρουσιάσω τις ίδιες προτάσεις και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας εύχομαι καλή παραμονή εδώ και καλές εργασίες. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι Θα ήθελα να ακούγεται πιο συχνά ότι η Ρουμανία χρειάζεται τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω και να την ακούσατε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Έλντερ Γκάρθια Θαμπάλ Ρουμπιάλ για την πρόταση κανονισμού για την θέσπιση του μηχανισμού προγραμμάτων στήριξης. Παρακαλώ, κυρία Κάρτια, θα μπαλέχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κύριε Έτιγκερ, καλή επιτυχία στη συνεδρίαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Καλημέρα σας, ε, κύριοι συμπρόεδροι. Όπως έλεγε και ο πρόεδρος Λιπεράτσκι, θέμα που μα απασχολεί σήμερα το πρωί είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ρόλος που διαδραματίζει στην συνοχή, στη σταθεροποίηση ε, και στη σύγκληση. Αυτός ο ρόλος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για αυτούς τους τομείς ε, που μας απασχολούν ήταν πολύ περιορισμένος μέχρι σήμερα. Στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν υπάρχουν εργαλεία που πραγματικά να λειτουργούν σταθεροποιητικά. Ούτε εργαλεία που μας ε, οδηγούν στη σύγκληση. Παρόλο που πολλής λόγος γίνεται για τη συνοχή, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Οι πολιτικές συνοχή ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη των πιο μειονεκτικών περιφερειών, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτό το ποιοτικό άλμα που έχουν κάνει στο παρελθόν και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Επομένως, γίνεται λόγος για πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Κοινοβούλιο στην αντιπρότασή του σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει ως βασική γραμμή εργασίας το εξή. Δεν μπορούμε να κόψουμε ούτε ένα ευρώ από την πολιτική συνεχή και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Η κρίση έχει αποδείξει ότι μια κοινή αγορά με ένα κοινό νόμισμα όπου δεν υπάρχει ολοκληρωμένη νομισματική πολιτική και δεν υπάρχει ε, ολοκληρωμένη φορολογική και δημοσιονομική ένωση, είναι μια Ευρώπη όπου υπάρχουν ε, αριθμίες. Και γι' αυτό οξύνονται οι αποκλήσει μεταξύ χωρών, μεταξύ περιφερειών και μεταξύ πολιτών εντός του ιδίου κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητεί να υπάρχει υπολογισμό στις ζώνες του ευρώ, να υπάρχει φορολογική δυνατότητα στη ζώνη του ευρώ. Ε, ε θέλουμε προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τα, τα συμμετρικά και τα ασύμετρα σόκα και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ. Όλα αυτά τα ζητάμε εδώ και χρόνια ως Κοινοβούλιο. Και το Συμβούλιο ποτέ δεν έχει συμφωνήσει σε καμία πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όμως ε, θα έλεγα ότι είναι ε, σε ευρυϊκό στάδιο αυτό που θα έπρεπε να είναι μια πραγματικά φορολογική ενιαία πολιτική και δημοσιονομική ε, πολιτική ενιαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή κάποια προκαταρκτικά βήματα πολύ πρόημα έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ το Συμβουλίο τα αρνείται όλα. Το πρόγραμμα στήριξη των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνεται στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. 25 δι θα δοθούν για να γίνουν διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη. Από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόταση αυτή παρόλο που η συζήτηση είναι ακόμα εν εξελίξη και υπάρχει ανταλλαγή ιδεών και γι' αυτό δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή πώς θα διαμορφωθεί η οριστική θέση μας. Ωστόσο, ε, κάνοντας ένα μικρό απολογισμό, μπορώ να σας πω για τα βασικά σημεία τη συζήτηση. Υποτίθεται ότι η πρόταση θέλει να λειτουργήσει ω κίνητρο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν εθνικέ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει όπω προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τα κράτη που είναι στο ευρώ και για να ενισχυθεί η σύγκληση με τι χώρε που θέλουν να προσχωρήσουν στο κοινό νόμισμα. Μπορεί τα 25 δις να φαίνονται σημαντικά, όμως για 27 χώρες και για 7 χρόνια είναι ένα ποσό πολύ περιορισμένο, πολύ μικρό παρόλο που ακούγεται μεγάλο και δεν θα οδηγήσει σε καμία μεταρρύθμιση. Και αν παραμένει η πρόταση έτσι όπως έχει, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, χάνεται στα μέσα της διαδρομής, γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για να ε, χρηματοδοτηθούν αυστηρά εθνικές πολιτικές. Το επαναστατικό θα ήταν να έχουμε μια αιρεσιμότητα, αλλά θετική αιρεσιμότητα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει να χρηματοδοτηθούν πολιτικέ οι οποίε κατοχυρώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά όντω οδηγούν στην επίτευξη των βασικών στρατηγικών που είναι η αηφόρος ανάπτυξη και η Συμφωνία των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως κράτη-μέλη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Άρα νόημα έχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση χρηματοδοτούμε, περιβαλλοντική, δημοσιονομική, του παραγωγικού τομέα, του εκπαιδευτικού συστήματος, να συνδέεται άρρηκτα με την επίτευξη αυτών των στόχων ε, πάνω στους οποίους ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε δεσμευτεί. Πολλής λόγος μπορεί να γίνει για το τι πρέπει και τι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και τι όχι. Σε κάθε περίπτωση να είμαστε ευέλικτοι και να μην κλείσει η πρόταση. Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της Ιρλανδίας που έλεγε ο Επίτροπος Έτιγκερ. Με το σκληρό Brexit η Ιρλανδία θα είναι από τις χώρες που θα πληγούν περισσότερο και αν χρειαστεί βοήθεια τότε δεν θα μπορεί μάλλον να, ε, χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στήριξη των μεταρρυθμίσεων, γιατί οι ανάγκε τη Ιρλανδία δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και άρα ή δεν μπορεί να το, χρησιμοποιήσει ή δεν μπορεί να περιμένει ότι οι ανάγκε τη Ιρλανδία θα συμπεριληφθούν στον επόμενο προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δηλαδή, Ανεξαρτήτως του κατά πόσο λέμε ότι η χή δέσμη μέτρων μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή όχι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Και αυτό είναι το βασικό σημείο των συζητήσεων που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το πρόγραμμα είναι επίσης σημαντικό διότι στηρίζει τις άμεσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και έχει μια γραμμή τεχνικής βοήθειας. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά αποτελεσματικό και αναγκαίο και γι' αυτό υπάρχει τεράστια ζήτηση από πλευράς χωρών για την γραμμή τεχνικής στήριξης και γι' αυτό έχει νόημα και είναι και λογικό να αυξηθεί το κομμάτι του προπολογισμού που δίνεται στην τεχνική βοήθεια. Και έχουμε και μια γραμμή του προπολογισμού που, για τις χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν στο ευρώ. Και πρέπει να πλαισιωθούν προς αυτή την κατεύθυνση γιατί γνωρίζουμε ότι το, τα χρήματα που έχουν επιμεριστεί για αυτές τις δράσεις είναι πολύ λίγα και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν αποφασιστικά, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια σημαντική βοήθεια, ειδικά αν αυξήσουμε το ύψος των διαθέσιμων ποσών. Τώρα, τα κριτήρια διανομή πρέπει να αναθεωρηθούν κατά τη γνώμη μα. Αυτή τη στιγμή βασίζονται μόνο στο πληθυσμιακό κριτήριο των χωρών και το ο πληθυσμό μπορεί να είναι αντικειμενικό κριτήριο, είναι όντω, αλλά δεν είναι επαρκέ. Δεν φτάνει από μόνο του ω κριτήριο. Σε σχέση με την ανάγκη και τη βούληση ενό κράτου να, προβεί σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Ο πληθυσμό δεν έχει σχέση με το κατά πόσο μπορεί το κράτο μέλο να χρηματοδοτήσει αυτέ τι μεταρρυθμίσει με ίδια μέσα. Μπορεί να έχει μεγάλο πληθυσμό δηλαδή και να μην μπορεί να τι χρηματοδοτήσει. Τέλος, η χρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων δεν λύνεται με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να το αλλάξουμε και να το ε, κάνουμε μια ευκαιρία έτσι ώστε τα ε, κράτη να δουλέψουν προς κοινού στόχους που θα ωφελήσουν τους πολίτες, δηλαδή στην κοινωνική σύγκληση, στη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αηφόρο ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και πάνω σε αυτές τις τάσεις και κατευθύνσεις εργαζόμαστε εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, όπω είπαμε. Δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα πέντε λεπτά. Έρχομαι στους επόμενους ομιλητές μας, που είναι η κυρία Περβάνς Μπερές και ο Χωσέ Μανώλη Φερνάντες, που είναι ευρωβουλευτές και εισηγητές της πρότασης για ένα κανονισμό για τη δημιουργία προγράμματος στήριξης μεταρρυθμίσεων. Κυρία Περβάνς Μπερές, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ρουμανική Προεδρία που προχωράει σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και όπου χρειαζόμαστε πραγματικά κάθε όθηση. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητοί πρόεδρε, είναι σημαντικό όταν εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές βρίσκονται μαζί. Ήμουνα υπάλληλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλλον διορθώνει η κυρία Μπερές, στην Γαλλική Εθνική ε, Συνέλευση με τον Λοράν Φαμπιούς όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα και αυτή η φορά είναι η τελευταία μου, οπότε καταλαβαίνετε για μένα έχει μεγάλη σημασία και συζητάμε για ένα θέμα που χρειάζεται από κοινού προσπάθεια από τις δύο πλευρές της νομιμότητας. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να επενθυμισω τέσσερις πέντε αρχές που για μένα είναι βασικές. 25 χρόνια λοιπόν είμαι ευρωβουλευτής και δουλεύω για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προπολογισμού, προπολογισμού της Ένωσης και φοβάμαι ότι τον Απρίλιο θα εγκαταλείψω τα καθήκοντά μου χωρίς να έχω πετύχει αυτό το στόχο. Πάντως κάποιοι το είπανε. Χρειάζεται ένας ειδικό προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Εγώ δεν θέλω να είναι η Ευρωζώνη ένα κλειστό όμιλο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μα παρόλα αυτά το τι σημαίνει να είναι κανεί μέλο στην Ευρωζώνη. Τα υπέρ και τα κατά. Και στα κατά υπάρχει και η εγκατάλειψη ή μεταφορά κάποιων περιθωρίων στο policy mixed σε βάρος των χωρών μελών. Όμως αυτή η μεταφορά δεν έγινε, γιατί είχαμε το ίδιο νόμισμα, χωρίς όμως να επωφεληθούμε και από μηχανισμούς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στις αντικυκλικές περιόδους. Και ακριβώς γι' αυτό πρέπει κάτι να αλλάξει την Ευρωζώνη. Δεύτερη αρχή. Πρέπει στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται και μας προβληματίζει. Εγώ απαντάω ναι και νομικά είναι εφικτό. Και αυτό κάναμε όταν ήμασταν ε, στο ανώτερο σημείο της ε, κρίσης και δημιουργήσαμε το MSF που ήταν ένας μηχανισμός προσαρμοσμένος στην κρίση και στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους που εγγυόταν ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως παρόλο που η κρίση ήταν στις χώρες της Ευρωζώνης και ακριβώς Γι' αυτό μας χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο. Τρίτον, έχουμε στο τραπέζι και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με μια λειτουργία σταθερότητας. Αποτελεί μια εμβριακή μορφή ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης. Είναι μια καλή πρόταση. Και λυπάμαι που το ζεύγο στο γαλλογερμανικό που συνήθως ηγείται αυτών των θεμάτων μας ξαναβάζει στους ψιλοκαυγάδες αντί να χτίσει πάνω σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής που είναι μεν μετριοπαθής αλλά που έχει να κάνει με τη βασική λειτουργία που χρειάζονται οι χώρες μέλη που δεν είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας που δεν αφορά μόνο τις χώρες ευρώ, που δεν είναι το θέμα της σύγκλησης έτσι όπως προτείνεται στα συμπεράσματα των χωρών της ζώνης του ευρώ και που δεν μιλάμε για ελλείμματα, αλλά είναι η λειτουργία της σταθερότητας, σταθεροποίησης. Και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια έκκληση, να σας ζητήσω ως εθνικοί βουλευτές να την κοιτάξετε προσεκτικά αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αγνοεί το Eurogroup και το Συμβούλιο σήμερα, ενώ αποτελεί ένα μέσο για να βγούμε από το διέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Χάμερ εκπονήσαμε μία βάση συμβιβασμού που μας επέτρεπε να χτίσουμε πάνω σε αυτό το βήμα, διευρύνοντας ε, τις δυνατότητες παρέμβασης που θα μπορούσαν να πρικοδοτήσουν αυτό τον ε, μηχανισμό υπέρ της ανεργίας, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της. Δυστυχώς όμως ε, δεν προχωρήσαμε. το ΕΛΚ παρετήθηκε, ο εισηγητής εκεί. Αν εσείς μπορείτε να κάνετε ε, πώς θα το να πιέσετε το ΕΛΚΑ να βάλει κάποιον άλλο θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ξέρω, σας ζητάω πολλά. Αλλά η δικιά σας κινητοποίηση για αυτήν την λειτουργία σταθεροποίησης είναι και το σημαντικό μήνυμα που θέλω να φέρω εδώ από αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χώσε Μανώλ Φερνάντος. Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εύχομαι τα καλύτερα στην ε, Προεδρία της Ρουμανίας. Καλώς ορίζω τους συναδέλφους ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αγαπητοί Περβάνς, δεν φταίει το ΕΛΚ. Το ΕΛΚ πάντα βρίσκει λύσεις ε, ενωτικές. Δεν, φταίει. δεν μπορεί να φταίει το ΕΛΚ αν δεν προχωράει η υπόθεση αυτή. Πρόκειται για μια πρόταση που απαιτεί μετριοπάθεια, στάθμιση λογική. Η αλληλεγγύη λοιπόν και η υπευθυνότητα σε σχέση με τις ε, υποσχέσεις που έχουν δοθεί είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, και πρέπει να σταθμιστούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα βήμα επιπλέον, ένα βήμα που γίνεται με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που πρέπει να ε, μελετήσουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται να δείξουν και το πνεύμα αυτό της πίστης τα, οι εθνικές κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο θεωρείται αυτονόητο, αυτό το πνεύμα πίστης, ε, μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Ταυτόχρονα αυτή η πίστη σημαίνει, ε, η αξιοπιστία σημαίνει να πληρούνται οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, προτάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά θα έπρεπε και ε, το Eurogroup, παραδείγματι, να έχει ένα σαφέστερο ρόλο. Ενώ δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει τίποτα για το Eurogroup για να προχωρήσει. Ε, θα ήταν επωφελής προς όλους βέβαια μια ευρωζώνη ισχυρή. θα είχαμε ένα εργαλείο προληπτικό με βάση την αρχή ότι είναι καλύτερο να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Και άρα με τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε μία εκτέλεση στην ευρωζώνη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που θα είχε και μια υποστήριξη μετά έχουμε το Ταμείο των Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΣΕ σχέδιο Juncker, το οποίο σε ορισμένε χώρε που έχουν μεγαλύτερε δυσκολίε μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Ε, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Εστονία και άλλε έχουν ωφεληθεί πολύ περισσότερο ε, σε λόγο ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν, μιλούμε για έναν ε, προϋπολογισμό με γραμμές ειδικέ αφιερωμένες στην Ευρωζώνη με πολύ συγκεκριμένα και είναι πολύ θετικό αυτό στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 30 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούμε να επαληθεύσουμε βεβαίω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να βρούμε μέσα που θα μας επιτρέπουν ταχεία αντίδραση, αυτόματη θα έλεγα αντίδραση, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα. Όσο προχωρημένη και είναι η ενοποίηση στο πολιτισμο οικονομικό πλαίσιο, να έχουμε ένα μέσο το οποίο θα μας επιτρέπει να αντλήσουμε τους απαραίτητους πόρους σε κατάσταση ανάγκης. Ένας μηχανισμός δηλαδή, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει τα πρώτα βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ε, αργότερα σε έναν ε, προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Αλλά πάντα θα υπάρχει ένας έλεγχος από το Ευρωπαϊκό... Αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει ένας, ένας έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι του ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην αποκλειστεί. Είναι κάτι το οποίο ε, απαιτείται. Γι' αυτό υποστηρίζουμε και την συνήθη νομοθετική διαδικασία μια διαδικασία καλή με χρήσιμα εργαλεία και πορεία και ελπίζω, ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει, ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα δείξει την ίδια φιλοδοξία, θα το πω έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το ρεαλισμό, γιατί δεν είναι μόνο φιλοδοξία, είναι και ρεαλισμός να αποδεχθεί αυτά τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία της Ευρωζώνης. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τον κύριο Εύερτ Γιάνν Σλότβεκ από το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητά μέλη της Ρουμανικής Προεδρίας, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου έδωσαν να αναπτύξω ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερο στα εθνικά κοινοβούλια, να παρουσιάσω τους στόχους του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα θέλαμε να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από δική μα πλευρά για την εξαιρετική του εργασία κατά τη διοργάνωση αυτή αυτή, αυτής πολύ σημαντική συνεδρίαση. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα τα Ολλανδικά. Σήμερα το πρωί και χτες μιλήσαμε πολύ για νέους στόχους και νέους μηχανισμούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη πιο συγκεκριμένα. Οικονομικά βέβαια υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη, άρα είναι κατάλληλη στιγμή για να φτιάξουμε, όπως λέμε, τη στέγη του σπιτιού μας τώρα που ο ήλιος λάμπει. Επίσης, σε αυτές τις συζητήσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να προσέχουμε τους μηχανισμούς και τους στόχους που ήδη διαθέτουμε. Σε αιτήσιο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού προειδοποίησε το νεκτικό συνέδριο τον Οκτώβριο που μας πέρασε ε, για το ότι έχουμε ένα ρεκόρ καθυστερημένων πληρωμών επειδή δεν είχαμε την προσφορά αρκετών ε, καλών ε, σχεδίων. Έτσι, έχουμε φτάσει σε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 267 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο έλεγχος επίσης προειδοποίησε και για μια κατάσταση όπου θα έχουμε υποσχεθεί υπερβολικά πολλά, τα οποία δεν θα μπορούμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, σήμερα μιλάμε για συνοχή, σταθεροποίηση και σύγκληση. Είναι πολύ καλό να λάβουμε υπόψη μας στη συζήτηση αυτή της προειδοποίησης του λεκτικού συνεδρίου και να φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους μηχανισμούς που ήδη διαθέτουμε. Εγώ θα τόνιζα το βασικό μέσο που διαθέτουμε για την συνοχή και τη σύγκληση που ήδη υπάρχει και που είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο μακροπρόθεσμος αυτός προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατεξοχήν ένας πολιτικός μηχανισμός ο οποίος μας βοηθάει πολύ να καλύψουμε τις προτεραιότητές μας. Πρέπει να κάνουμε βέβαια επιλογές και να θέσουμε προτεραιότητες συγκεκριμένα, γιατί το κάθε ευρώ μία μόνο φορά μπορεί να ταπανηθεί. Για το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, λοιπόν, υπάρχουν τρία θέματα που μα απασχολούν. Εμεί θέλουμε έναν αποτελεσματικό προπολογισμό, έναν υπεύθυνο προπολογισμό και ένα σύγχρονο προπολογισμό. Εδώ θα σας μιλήσω για κάθε ένα από τα τρία αυτά στοιχεία για να σας παρουσιάσω τις απόψεις του Ολλανδικού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον στόχο σταθεροποίησης της Οικονομικής και Νομισματικής ε, Ένωσης. Πρώτα απ' όλα για αποτελεσματικό προπολογισμό. Α αρχίσουμε με τον Brexit. Το Brexit εννοείται ότι είναι κάτι δυσάρεστο και θα κάνει μεγάλη ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στην Ολλανδική οικονομία, η οποία είναι μία από αυτές που θα χτυπηθούν περισσότερο μετά το Brexit. Συγχρόνως, οι κάτω χώρε είναι και ένας από τους βασικούς καθαρούς εισφορείς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώ μα αναγκάζει το Brexit να ξανασκεφτούμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και συγχρόνω όμω να δούμε Ποιε είναι και ευκαιρίε που μα δίνει και μεταρρυθμίσει. Οι περισσότεροι στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, λοιπόν, θέλουν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να αντικατοπτρίζει την ε, μείωση που θα έχουμε λόγω του ότι από 28 θα γίνουμε 27. Με τη στήριξη λοιπόν της πλειοψηφίας του Ολλανδικού Κοινοβουλίου εμείς λέμε ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να μειωθεί να παραμείνει το ίδιο, όπως και πριν την αποχώρηση. Γιατί αλλιώς θα πρέπει δυσανάλογα να πληρώνει η Ολλανδία. Δεύτερον, υπεύθυνο προπολογισμό. Για μας είναι κάτι πολύ βασικό αυτό για τις δαπάνες για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη βάση της κοινωνίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πολίτης να γνωρίζει ότι τα χρήματα που πληρώνει με τους φόρους ξοδεύονται καλά. Γι' αυτό ζητάμε από όλες τις χώρες μέλη να κάνουν το ίδιο που κάνει και η Ολλανδία, δηλαδή να διαχειρίζονται καλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να ετοιμάζουν και δηλώσεις όσον αφορά τη διαχείριση των ενισχύσεων αυτών με διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ένας καλός έλεγχος και αυτός γίνεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Η αρχή της χρηματοδότησης ε, να ελέγχεται, όπως επίσης να αξιολογούνται και οι δαπάνες. Πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία για κάθε κονδύλιο που δαπανούμε. Έτσι μόνο θα, περάσουμε, ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να βοηθήσει ε, τους ανθρώπους που ζουν και σε νοσιακές περιοχές να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Έπειτα, σύγχρονος προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί ότι η συνοχή και η σύγκληση των οικονομιών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό χρειάζεται εξυγχρονισμός του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι επίσης σημαντικό και για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μια σταθερή ευρωζώνη απαιτεί οι, χώρες μέλη να κάνουν και τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έπειτα, πρέπει να στηρίξουμε οικονομίες αντοχής και αυτό βέβαια το κάνουν οι χώρες μέλη. Όμως ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό και το Ολλανδικό Κοινοβούλιο θέλει θετικά κίνητρα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό υπέρ μεταρρυθμίσεων. Και θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Οι διαφορετικέ λοιπόν μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν στι χώρε μέλη έτσι όπω αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυτή είναι στόχη που στηρίζει η πλειοψηφία του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θέλουμε ένα εξυγχρονισμένο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που μπορεί πολλά να προσφέρει. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής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 για την Ευρώπη της σύγκλησης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και θέλω να το τονίσω στην πρώτη μου παρέμβαση. Εγώ είμαι πεπισμένος ευρωπαϊστής, ξέρετε. Θυμάμαι ότι έχω από πολύ νωρίς προσχωρήσει στις αξίες των ιδρυτών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προσχώρηση της Πορτογαλίας το 86, με την πτώση του τείχου στο Βερολίνο, με το άνοιγμα προς τα Ανατολικά, με την ε, ε, προσχώρησή μας στο ευρώ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στάδια και όλοι οι νέοι της εποχής μου συμμερίζονταν αυτό το ευρωπαϊκό ιδανικό. Δυστυχώς όμως σήμερα η πραγματικότητα αυτή έχει αλλάξει άρδιν. Πολλοί πια δεν πιστεύουν στο ευρωπαϊκό όνειρο ούτε στο ευρωπαϊκό όραμα και θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προκειμένου να ξαναπάρει τα πάνω του το ευρωπαϊκό εγχείρημα κάτι πρέπει να αλλάξει. Και ένα από τα εργαλεία που έχουμε για να επιφέρουμε αυτές τις θετικές αλλαγές είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Έχουμε θετικές προτάσεις ε, στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλει να ενισχύσει τους ίδιους πόρους, θέλει να ενισχύσει ε, τον εξοχρονισμό του προϋπολογισμού στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφοριακής οικονομίας, τη καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής του καλύτερου ελέγχου των συνόρων των προγραμμάτων στήριξης της νεολαίας. Θέλει θετικό προπολογισμό για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, για καλύτερη και περισσότερη διαφάνεια, για ανάληψη ευθυνών με χάρη ε, για ανάληψη ευθυνών χάρη στο καλύτερο έλεγχο και την καλύτερη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη σύγκληση, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις σχέσεις που θα μας επιτρέψουν να κινητοποιήσουμε δημόσια κονδύλια και ιδιωτικά. Απλούστευση, ε, βελτίωση της διαδικασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύτερη προσαρμογή των προγραμμάτων στην πραγματικότητα. Όλα αυτά επιθυμούμε, όλα αυτά ε, ε, επιδιώκουμε, γιατί η πραγματικότητα σε κάθε χώρα μπορεί να είναι διαφορετική και δεν θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο να βασιζόμαστε στο βαθμό εκτέλεσης του προπολογισμού και στο βαθμό χρήσης των δαπανών. Είναι θετικά λοιπόν όλα αυτά. Η πρόταση όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την Πορτογαλική κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και συμφωνώ με την επίσημη θέση της χώρας μου. Και γι' αυτό χαιρετίζω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε οι νέες πολιτικές να αναπτύσσονται χωρίς να θέτουν σε αμφισβήτηση τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό για υφιστάμενα προγράμματα και για τη σύγκληση και τη συνοχή η σύγκληση είχε προβλεφθεί ως μία από τις βασικές αρχές στη συνθήκη της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1957. Και για η σύγκληση είναι προϋπόθεση για να μιλήσουμε για την επιβίωση του ευρώ και να μην το αφισβητήσετε αυτό κυρίες και κύριοι. Το ευρώ θα επιζήσει και θα επιβιώσει και θα πάει μπροστά μόνο αν έχουμε συνοχή στην Ευρώπη που να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση και που να πλησιάζει όλο και περισσότερο ο ένας τον άλλον. Η σύγκληση λοιπόν είναι θεμελιώδες ε, στοιχείο για να έχουμε τη στήριξη των λαών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ε, Εάν θέλουμε μια Ευρώπη που να βασίζεται στη στήριξη των πολιτών της, τότε θα πρέπει όλοι να έχουν θετική εικόνα, να έχουν εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η σύγκληση είναι κάτι το θετικό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάποιες χώρες γιατί ε, ε, ωφελούνται από την καλή διαχείριση των οικονομιών τους, αλλά η σύγκληση είναι καλή και για τις άλλες χώρες γιατί έχουν περισσότερα κέρδη. Αν, έχουμε μια εσωτερική αγορά πιο ισχυρή και με μεγαλύτερη συνοχή, τότε και οι ισχυρές χώρες έχουν περισσότερα κέρδη. Και θα έλεγα ότι κάθε ένας από εμά πρέπει να κάνει το ό,τι μπορεί για να καλλιεργήσει στο Εθνικό του Κοινοβούλιο τη στήριξη στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα Εθνικά Κοινοβούλια να ενισχύσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητεί την ενίσχυση του κοινοτικού προπολογισμού. Η Πορτογαλία ήδη το έχει δηλώσει αυτό και πρέπει να το κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε νέε πολιτικέ να αναπτύσσονται χωρί να θέτουν σε κίνδυνο τι παραδοσιακέ μα πολιτικέ. Και τέλο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα ένα τελευταίο προβληματισμό που ανέφερε και ο Επίτροπος Έτιγκερ. Η σημασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Καθυστερήσεις έχουμε εκεί. Για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την εξηγίαση των τραπεζών και για την εγγύηση των αποταμιεύσεων. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα δυναμικό που να στηρίζεται στην ενίσχυση των πολιτών, στην αποδοχή των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιπρόεδρος Λιμπεράτσκι έχει το λόγο για να κατευθύνει τις συζητήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Μιχαλέψου. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο αυτό που μας δώσατε με τις ομιλίες σας. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τον χρόνο για τη συζήτηση. Βλέπετε τις θέσεις του Κοινοβουλίου αφενός, της Επιτροπής Αφετέρου, κάποιες παρατηρήσεις που εκπροσωπούν στο Συμβούλιο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Με την αδειά λοιπόν θα γυρίσω και εγώ στην μητρική μου γλώσσα τα πολωνικά. Καταρχάς λοιπόν θα ακούσουμε τον κύριο από την ε, Ρουμανία, πάλι ε, Ένα λεπτό όμως, επειδή έχω, <laughs> ξέρετε, μακρά πείρα και είμαι γνωστό ότι κλείνω τα μικρόφωνα όταν κανεί μακρηγορεί. Να έχετε και το νου σα. Κύριο Κόκου, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια γνήσια συζήτηση για το μελλοντικό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο από την περίοδο 2020 και μετά. Μία αγνήσια συζήτηση που θα εξασφαλίσει την σύγκληση και τη σταθερότητα στην Ευρώπη πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορες ε, διαστάσεις, διάφορα θέματα και βεβαίως θα πρέπει να ε, εκτίθεται στο δημοκρατικό έλεγχο από πλευρά των πολιτών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω και εγώ δύο λόγια για την πατρίδα μου, τη Ρουμανία. Είναι πολύ σημαντικές ε, για μας οι δομές, τα ποσά, τα κονδύλια που θα στηρίξουν την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό θα είναι άλλωστε και η εγγύηση της επιτυχίας της παρουσίας και της συμμετοχής της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τροφοδοτηθεί ο λαϊκισμός και οι αντιευρωπαϊστές. Συγκεκριμένα τώρα, επιτρέψτε μου να επισημάνω τα εξής. Η πολιτική της συνοχής πρέπει να παραμείνει σε ένα χωριστό κεφάλαιο. Πρέπει οι συνοριακές διαστάσεις ε, να προβληθούν ιδιαίτερως με στόχο την περιφερειακή και οικονομική συνοχή μέσα στην ίδια περιφέρεια πέραν των εθνικών συνόρων. Πρέπει να προωθηθούν ε, νέα εργαλεία για το προσεχές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με λύσεις οι οποίες θα λύσουν και τα προβλήματα στον προπολογισμό το σχετικό με την έρευνα, στην, ε, ε, στις άμεσες πληρωμές και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου προσφέρατε να σας παρουσιάσω τις θέσεις μου εκ μέρους των συναδέλφων του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Να, μας εξασφαλίσατε και έξι επιπλέον δευτερόλεπτα στον περιορισμένο κοινοβουλευτικό χρόνο. Πολύτιμα. Μια και τελειώσατε λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Μπάχα από τη Γερμανία, πρόεδρε. Φρονώ πως βρισκόμαστε ενώπιον θεμελιωδέστατων προκλήσεων εμείς στην Ευρώπη Δεν λειτουργούν πλέον τα παγκόσμια σταθεροποιητικά συστήματα. Δεν επαρκούν, δεν είναι πια δυνατό να διατηρηθεί με τόση ευκολία η συνοχή της Ευρώπης. Το Brexit έρχεται χωρίς να είναι δυνατόν κανείς να προβλέψει τον ευρύτερο αντίκτυπο και τις συνέπειές του. Βλέπουμε μια πολιτική διχασμού και κατακαιρματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα τίνουν ε, στην, ε, στον καταμερισμό, στο διαμήρασμα του κόσμου και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε μόνο από κοινού να εξασφαλίσουμε για την ευρωπαϊκή οικονομία την προστασία της έτσι ώστε να μην χαθεί έναντι των Ευρωπαίων, ε, των Αμερικανών βιομηχανικών γιγάντων αφενός και των Κινέζων ψηφιακών μεγάλων αφετέρου. Όλα αυτά είναι οι προκλήσεις της εποχής μας. Πρέπει τη σύγκληση λοιπόν να την προσφέρει μαζί με μια λύση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα προχωρήσει σε έγκριση. Έχουμε ένα μεγάλο πλεόνασμα στον γερμανικό προϋπολογισμό, ωστόσο πρέπει να δώσουμε έμφαση και στο εμπορικό έλλειμμα που υπάρχει σε σχέση συγκεκριμένα με τους ψηφιακούς γίγαντες μέχρι και 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τους Αμερικανούς ψηφιακούς γίγαντες. Έτσι λοιπόν αυτά όλα πρέπει να μπουν στην πλάστιγκα και να ε, εξασφαλίσουμε μια πιο δίκαιη κατανομή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να έχουμε έναν ε, προϋπολογισμό της Ευρωζώνης που θα είναι αποδεκτός από όλους και για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Πάλι σας ευχαριστώ βεβαίως που σεβαστήκατε το, λόγο, το χρόνο σας. Ο κύριος Μάρτας για την Ελλάδα, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά. πολιετέ δημοσιονομικό μα πλαίσιο τη περίοδου 2021-2027, εκτό από το σκέλο των δαπανών, θα ήταν σκόπιμο ενδεχομένω να εξεταστούν και νέοι πόροι εσόδων. Και αυτό έχοντα υπόψη και τον Brexit. Ένα νέο πόρο στον προπολογισμό τη Ένωση θα μπορούσε να προκύψει από τα ακόλουθα. Αναλυτικότερα ο κανονισμός 1176-2011, ε, που είναι ο πέμπτος κανονισμός από το πακέτο των έξι μέτρων, συνδέει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και με τα ισχυρά πλεονάσματα του ισοζυγίου των τροξών συναλλαγών λόγου χάρη. Αντίθετα, οι άλλοι τέσσερις κανονισμοί και μία οδηγία των έξι μέτρων, του πακέτου των 6 μέτρων, συνδέουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες με τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Έχοντας υπόψη ότι τα εμπορικά υπερπλεονάσματα είναι το προϊόν και της ανοιχτής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου κάποια κράτη-μέλη αντλούν ιδιαίτερα πολλά ωφέλη, τότε θα μπορούσε να προβλεφθεί το εξή. Κράτη-μέλη που καταγράφουν πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών άνω του 4% του ΑΕΠ, παραδείγματο χάρη, θα μεταφέρουν τα υπερπλεονάσματά του στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιούνται είτε για να καλύψουν ανάγκε ενιαία πολιτική είτε για να βελτιώσουν τη ρευστότητα στην αγορά κρατών μελών που επιδιώκουν να εκπληρώσουν τους στόχους που προβλέπονται στο πακέτο των δύο μέτρων και στο δημοσιονομικό σύμφωνο. Στο πλαίσιο όλα αυτά, στο πλαίσιο των προσπαθειών για σύγκληση και συνοχή στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you very much. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριος Μάιστοβιτς, ε, Πολωνία. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει και γι' αυτό θα περιοριστώ μόνο σε ορισμένα από τα σχόλια που ακούστηκαν και πολύ γενικά. Ε, Βεβαίω και είναι αυτονόητο όσο περισσότερε είναι οι χώρε που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη να υπάρχει και περισσότερο Κέρδο και όφελο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και την Ευρωζώνη συνολικά. Εδώ λοιπόν η Πολωνία βρίσκεται σε μια ιδιάζουσα κατάσταση γιατί ναι, έχουμε προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή Συνθήκη η οποία αναφέρεται στην ε, ένταξη στην Ευρωζώνη αλλά χρονοδιάγραμμα δεν έχει προβλεφθεί και δυστυχώς για την Πολωνία αυτό θα σήμαινε και σταγματική αλλαγή για έγκριση από το Εθνικό Κοινοβούλιο Πράγμα το οποίο θα ήταν ε, μάλλον δύσκολο να εξασφαλιστεί και ε, το παράδειγμα της Σλοβακίας αλλά και άλλων κρατών που πρόσφατα έχουν υιοθετήσει το ευρώ ε, δείχνει ότι ανεξάρτητος του αν η οικονομία είναι σε καλή ή κακή κατάσταση την ώρα που εισάγεται το νόμισμα η έκβαση δηλαδή ο αντίκτυπος από την εισαγωγή του κοινού νομίσματος ήταν πάντα θετικός. Η Πολωνία, η πολλές πολιτικές ε, ομάδες και οικογένειες της Πολωνίας έχουν καταστήσει προτεραιότητά τους ε, και την ανταξη Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν και στην Ευρωζώνη τώρα. Εμείς είμαστε μια από αυτές και πρέπει να επιταχυνθεί αυτό το βήμα. Η κατάρτιση ενός χωριστού προϋπολογισμού για την Ευρωζώνη επίσης θεωρώ ότι μπορεί να έχει θετικό αλλά και, αλλά και αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαμε ως εθνική οικονομία δηλαδή να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση των οικονομικών αποφάσεων αλλά και των καταστάσεων των οικονομικών εάν ήμασταν μέλος της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι και το επιχείρημα των πολυάριθμων ευρωσκεπτιστών που ε, όλο και τώρα μιλούν ε, κατά της Ευρώπης και της Ευρωζώνης τελευταίο καιρό, θα μπορούσαν δηλαδή αυτοί οι ευρωσκεπτικιστές να πιέζουν για να παραμένει πάντα στο περιθώριο της Ευρωζώνης ε, η Πολωνία. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να πράξουμε θα είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ε, κάνουμε την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την πληροφόρηση που χρειάζεται για τη σημασία της Ευρωζώνης, όχι μόνο για τις οικονομίες αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα. Τα νοικοκυριά να δουν ότι τα συμφέρει η ε, ένταξη στην Ευρωζώνη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πορτογαλία, πες. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Μαρκές. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να αποτελέσει το μέσο σύγκλησης, σταθεροποίηση και συνοχής. Αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε επίσης τα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν με τη στρατηγική της Λισαβόνα και όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης που τονίζουν ότι τελικά η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά ευάλωτη και δεν θα έπρεπε να συνδυαστεί με ένα χρηματοδοτικό μέσο, με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να πάρουμε και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δίχως άλλο, πρέπει να χρησιμεύσει για τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα για τους στόχους που έχουν να κάνουν με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θυμάμαι και μάλλον υπενθυμίζω αντιμετώπιση των ασυμμετριών, των ε, σοκ, των ασυμμετρικών ε, κλπ. Τα λόγια όμως πρέπει να γίνονται πράξη, να υπάρχει πραγματικά στήριξη στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν βλέπουμε την μείωση των ποσών στην πολιτική συνοχής, για παράδειγμα, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε ότι τελικά οι στόχοι αυτοί δεν υλοποιούνται, δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτό που ενέκρινε στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα είναι πολύ καλό για να αντιμετωπιστούν ακριβώ αυτέ οι περικοπέ και κατά των μέτρων μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Θέλω όμω να υπογραμμίσω ε, δύο πράγματα ακόμα από την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Μέσο Σταθεροποίησης υπέρ των επενδύσεων. Είναι ζωτική σημασία στο μέσο αυτό να αποτελέσει ένα γερό μέσο, ένα γερό μηχανισμό. Και δεύτερον, αυτό το παράθυρο που ανοίγει για τη δημιουργία ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης. Ξέρω ότι έχω περάσει το χρόνο μου, οπότε το μόνο που θα κάνω είναι θα επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Περβάνς. Αυτό ήθελα να κάνω, αλλά δεν έχω χρόνο, οπότε αρκούμε σε αυτά που είπε εκείνη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπός έχει το λόγο από την Ουγγαρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ σε ένα θέμα το οποίο ίσως δεν προσέξαμε αρκετά σήμερα αλλά είναι αναπόφευκτο να μιλήσουμε γι' αυτό. Και είναι η θέση των Υπουργών Οικονομικών. Η ναι θα ενισχυθεί και θα είναι ένα σημαντικό βήμα όταν έχουμε μια κοινή νοοτροπία μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ο ένας λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών είπε πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες για χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Θα εμβαθύνει ο λόγος του το χάσμα μεταξύ των χωρών μελών και θα υπονομεύσει ολόκληρη την κοινότητα. Εμείς πρέπει να συνυπάρχουμε μέσα σε νομιογενές πλαίσιο. Αν υπάρχουν χώρες οι οποίες θα μείνουν στην περιφέρεια Ισαΐ χωρίς βοήθεια, τότε θα υποφέρει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη θα μείνει πίσω όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι αυτή η θέση ενός Υπουργού Οικονομικών δεν είναι σωστή και δεν βοηθάει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Φαγαμάκη, η Φιλανδία. Παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γενικά μιλώντας, το επίπεδο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να ευθυγραμμίζεται όσο γίνεται περισσότερο με τα επίπεδα του GNI. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αύξηση, διότι πολύ λίγες χώρες έχουν υψηλότερη συνεισφορά. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να λάβουμε υπόψη μας όλες τις ε, πτυχές, γεωργία κλπ. Πρέπει επίσης να εγκρίνουμε έκτακτες δαπάνες μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό να επικεντρωθούμε στην καινοτομία και σε άλλους τομείς και θεωρούμε ότι περισσότερη ευελιξία χρειάζεται στο μέλλον. Τώρα το διοικητικό άχθος επίσης θα πρέπει να μειωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Όταν δίνονται κονδύλια θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι το πλαίσιο θα πρέπει να είναι επίσης περισσότερο προβλέψιμο, κυρίως στο τέλος της προγραμματικής περίοδου. Η πολιτική συνοχή τώρα. Οι εθνικές αρμοδιότητες και η ευθύνη των χωρών μελών θα πρέπει να διατηρηθούν με εργασιακές μεταρρυθμίσεις, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις κτλ. Και πιστεύουμε ότι είναι καλή η πρόταση της Επιτροπής αυτό, γιατί στηρίζει προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την υλοποίηση των ειδικών αναχώρασης στάσεων σε αυτές. και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Το καλύτερο πράγμα για να υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά είναι η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να δούμε την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κάτι γι' αυτό και να υπάρχει μόνιμη στήριξη για την Βόρεια και την Ανατολική Φιλανδία. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρότεινα να προβληματιστούμε πάνω στο ερώτημα της κυρίας Περβάος Μπερές. Αν χρειάζεται ειδικός προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα ήθελα να αναπτύξω στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Να σας υπενθυμίσω ότι στο αρχικό πρόγραμμα της δεκαετίας του 90 μία αγορά, ένα νόμισμα, η λειτουργία της σταθεροποίησης και της σταθερότητας εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Άρα, ε, πρώτη σκέψη είναι η εξή. Από τη στιγμή που σήμερα συζητούμε για ένα κοινοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ασύμετρων σοκ, τότε αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα κράτη της ζώνης του ευρώ έχουν παρετηθεί από ένα σημαντικό εργαλείο που είναι η ευελιξία ε, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το οποίο είχε το θάρρος να παραδεχτεί η κυρία Περβάν Μπερές, αλλά σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα και με τους κανόνες, τους δημοσιονομικούς που ε, ε, εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να βρουν τον απαραίτητο χώρο για να αντιμετωπίσουν τα ασύμετρα σοκ στην οικονομία τους. Έγινε λόγος για την αντίσταση του Eurogroup ο κύριος Φερναντές το είπε. Εγώ πιστεύω ότι το Eurogroup είναι ένας σκοτεινός μηχανισμός λήψης αποφάσεων που δημιουργεί προβλήματα δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται ακριβώς εκεί μέσα. Και Πρέπει να θυμηθεί κανεί ότι το Eurogroup γεννήθηκε ω αντιστάθμισμα στην ισχύ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θέλησε να είναι ένα πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα για να, έχουμε, να φτάσουμε στη θέση ενό Υπουργού Οικονομικών τη ζώνη του ευρώ, κάτι το οποίο ανέκαθεν ήθελε η Γαλλία. Και μετά την κρίση του ευρώ, το Eurogroup ήταν το εργαλείο αυτή τη διακυβερνητική προσέγγισης, την οποία έχουμε επανειλημμένω εδώ ε, υπογραμμίσει ε, και θεωρούμε ότι είναι ε, προβληματική και θα πρέπει αντίστοιχα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, καταλάβει πολύ περισσότερο χώρο και να έρθει στο προσκήνιο. Τα δύο θέματα αυτά σχετίζονται δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάχτα από την Πολωνία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολωνική προτεραιότητα ήταν ανέκαθεν πάντοτε η, η διαφάνεια και η ανοιχτή στάση σε αυτό το εγχείρημα της εμβάθυσης της νομισματικής ένωσης, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες, χώρες που σήμερα είναι εκτός Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη σύγκληση, με, τη σύγκληση με δύο τρόπους, μέσω του προϋπολογισμού, μέσω των περιφερειακών και διαρθρωτικών πολιτικών και μέσω του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Κυρίως όλα αυτά ως μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. στα θέματα σύγκλησης προς το ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος της, ε, του διαμοιρασμού των ευθυνών έτσι ώστε να χάνονται τελικά οι ευθύνες. Η Πολωνία πιστεύει ότι την ευθύνη για τη σύγκληση θα πρέπει να την έχουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που έχουν προσχωρήσει στο ευρώ, αλλά και τα κράτη-μέλη που έχουν επιλέξει να μείνουν εκτός ευρωζώνης. Εμείς πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε, ε, καταρχήν, ως αρχή, να είναι εργαλείο για να εγγυόμαστε τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών ανεξαρτήτως του συναλλάγματος, αν θέλετε, του νομίσματος που υιοθετεί το κάθε ένα από αυτά τα κρατημέλη. Άρα η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής με τα εργαλεία της έχει ως στόχο να αντισταθμίσει τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών και άρα αυτό πρέπει να παραμείνει ως βασικό εργαλείο ε, που θα χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε σύγκληση σε επίπεδο κρατών μελών. Σε αυτό το στάδιο της ευρωπαϊκής ελοκληρώσης η Πολωνία δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ και άρα δεν μπορεί να στηρίξει προτάσεις που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρόταση ενός ειδικού εργαλείου για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ Ω εργαλείο που θα πρέπει να περιληφθεί στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι η πρόταση της 14 η Δεκεμβρίου του 2018. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες μετά τις ευρωεκλογέ. Κατά τη γνώμη μας, ένα τέτοιο εργαλείο, εάν τελικά ήταν διαθέσιμο μόνο για τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στο ευρώ, μπορεί τελικά να αποδυναμώσει άλλε πολιτικέ και την γενικότερη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέτου από τη Ρουμανία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ήδη κατά τη συνεδρίαση Κόζακ των ε, Προέδρων στη Ρουμανία ε, οργανώσει συζήτηση με ακριβώς το ίδιο θέμα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω και τα συμπεράσματα της συνεδρίας αυτής της Κόζακ. Αγαπητοί φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνενώνει τις ε, δημοκρατικές κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών. Η λειτουργία η ίδια ενός δημοκρατικού κράτους θεωρείται προϋπόθεση για να προσφέρεται στον πολίτη το δημόσιο αγαθό, το βασικό δημόσιο αγαθό. Χωρίς αυτό λοιπόν ε, ζημιώνεται η κοινωνική συνοχή. Το κοινωνικό κεφάλαιο, ο κοινωνικός ιστός καταστρέφονται. Όταν η ανισότητα ξεπερνά το όριο αυτού που θεωρεί ως αποδεκτό ο πολίτης, όταν λησμονείται η κοινωνική δικαιοσύνη, η, ισοτιμία κινδυνεύει, η ισονομία κινδυνεύει η ίδια η δημοκρατία. Αυτό εξηγεί και την απώλεια κύρους και γοήτρου για το ευρωπαϊκό εγχείρημα που βλέπουμε να αμφισβητείται σε πολλά κράτη-μέλη. Χρειάζονται λοιπόν πολύ πιο ανοιχτές και περιεκτικές πολιτικές. Υπάρχουν ε, χώρες όπως η Ρουμανία που λόγω των χαμηλών μισθών, μισθών αλλά και της μεγάλης ανισότητας έχουν αντιμετωπίσει τεράστια διαρροή ε, ανθρώπων, εγκεφάλων όπως λέμε. Το Brexit, τεράστιο πλήγμα και για τις δύο πλευρές. Και Ίσα ίσα τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι συνέπειέ του και τα διδάγματα που πρέπει να αποκομίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια αναδιαμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό παραδέχονται πολλοί και είναι η πρώτη φορά ενδεχομένω που το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκινάει χωρί μια νέα στρατηγική. Χωρί μια στρατηγική όπω ήταν η στρατηγική τη Λιζαβόνας ή όπως ήταν η στρατηγική του 2020 τότε. Ε, δηλαδή φαίνεται να έχουμε μια ε, προσέγγιση ότι όλα πάνε καλά, συνεχίζουμε όπως πριν. Κι όμως δεν είναι έτσι. Είναι ένα υπόδειγμα δημιουργίας οικοδόμησης διεθνικής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε το δάσος όταν κοιτάμε τα δέντρα. Δεν πρέπει να... Ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ να ολοκληρώνετε την ανάγνωση. Το σύστημα των επιστροφών στη συμμετοχή στον προπολογισμό ορισμένων κρατών ε, καθαρών χορηγών δείχνει αυτή την ε, θεώρηση την, ε, της, του εθνικού κέρδους έναντι του κοινού ωφέλους. Υπάρχουν πολλά κράτη που υποστηρίζουν την κατάργηση αυτών των ειδικών ρυθμίσεων. Κυρία Κρέτσου, σας παρακαλώ, ναι, να τελειώσω. Και, και πρέπει να υπάρχει η λογική ενός ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού μέσα σε μια ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ θερμά, λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ιταλία παρακαλώ. Δυστυχώ το όνομα δεν το ακούσαμε. Στα αγγλικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Στα ιταλικά. Κατόπιν της ε, τελευταίας ε, παρέμβασης που άκουσα, θα ήθελα ιδιαίτερα να δώσω έμφαση στην ε, τελευταία αυτή πτυχή, δηλαδή τα προβλήματα που είχε άλλωστε και η τελευταία Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει και δεν κατάφερε να πράξει, δηλαδή την ενοποίηση των οικονομικών με τις κοινωνικές πολιτικές, το συγκέρασμα αυτών. Έγινε λόγος για συνοχή, για σύγκληση κτλ. σήμερα το πρωί. Αυτή όμως η συνοχή και η σύγκληση φοβούμε δεν εκφράζεται μέσα από κοινωνικέ πολιτικέ. Αυτή άλλωστε είναι και μια, ανισό, ε, μια συνέπεια την οποία είδαμε να εκδηλώνει και η τελική κυβέρνηση στην τελευταία της θητεία, τελευταία θητεία. Δηλαδή πίεσε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιταλική κυβέρνηση ε, να σταματήσει τα κοινωνικά μέτρα και αυτό οδήγησε σε αύξηση και της ενεργείας και βέβαια πολύ μεγάλη απογοήτευση για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των αγορητών εκ μέρου των εθνικών κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, εδώ στο Προεδρείο να δώσουν τις απαντήσεις τους πολύ σύντομα. Με ένα λεπτό το πολύ σας παρακαλώ να δώσετε τις απαντήσεις. Και ξεκινώ αντίστροφα με τον κύριο Ντουάρτε Πασέκο. Presidente, caros colegas, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, από τις διάφορες παρεμβάσεις νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο εξή συμπέρασμα. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των εθνικών ε, βουλευτών και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη θέση σας στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι θετικό, γιατί έτσι θα έχουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σλότβακ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κι εγώ ευχαριστήθηκα ακούσα και καταλαβαίνω ότι όλοι σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή, μια δυνατή Ευρώπη και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ενισχύσουμε επίσης την ανταγωνιστική δύναμη της Ευρώπης. Έχουμε να κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα και αυτό σημαίνει ότι το στο συνομικό πλαίσιο μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστική μας δύναμη και να προσφέρει όμως η και μια περισσότερο αλληλέγγυα Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα η υπερβάμωση έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ συγκρατώ από την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε τέσσερα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα το είπε και ο Μιχάλ Πακλαδί ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο όπου η Ευρώπη είναι μόνη της, οπότε μπορεί να είναι θύμα επιθέσεων. Με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι πολύ βασικό. Και άκουσα τι είπε η κυρία Μάρκες, ε, η φίλη από την Πορτογαλία αλλά και η κυρία Κρετού. Ναι, έχουμε μία νέα στρατηγική με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτή είναι η οικολογική διάσταση. Τουλάχιστον αυτό λένε οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε μαζί με άλλου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό μου προσφέρει μια κατευθυντήρια γραμμή στην Ευρώπη ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Όμω συγχρόνω δεν μπορούμε να μιλάμε για το διεθνέ πλαίσιο και για το Brexit χωρί να μετράμε πόσο πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη και πόσο χρειάζεται ένας αυτόματος σταθεροποιητής που να δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, μέσα σε Ευρωζώνης ανοιχτή σε όλους, χωρίς να μπαίνει εδώ ηθική διάσταση. Λυπάμαι που δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ήδη για την είσοδο στην Ευρωζώνη των χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμα και πιστεύω ότι μετά το Brexit αυτό θα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Έπειτα, για τη λειτουργία της σταθεροποίησης, δεν μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται μόνο στη διαιτησία των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών, γιατί υπάρχει και μια δυναμική στην Ευρωζώνη, η οποία απαιτεί έναν μηχανισμό αντιστάθμισης ή τέλος πάντων ε, άμβλησης των οικονομικών ε, αναταράξεων. Μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Μανώλη Φερνάντες τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα από τη δικιά μου τη πλευρά να πω ότι το κόστος είναι μεγάλο για την αντιμετώπιση των στόχων και κυρίως αν δεν έχουμε τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Το ότι δεν είχαμε μηχανισμό σταθερότητας, πόσο κόστισε στους Ευρωπαίους πολίτες η κρίση που δεν υπήρχαν ε, επίσης πόροι για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές και κάθε φορά να ψάχνουμε ειδικά ταμεία και καταπιστευτικούς μηχανισμούς για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Αυτό δεν βοηθά. Γιατί να συνεχίσουμε με αυτή την υποκρισία και να μην βρούμε τα κατάλληλα μέσα που χρειαζόμαστε. Έπειτα, δεύτερη παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία. Δεν ξέρω καμία χώρα μέλος που να έχει προπολογισμού όπου μόνο το 7% του προπολογισμού να πηγαίνει σε τρέχουσε δαπάνε. Σε κανένα προπολογισμό δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε όλοι αυτοί που μιλούν για τη μείωση των διοικητικών δαπανών, με αυτό έχει επιπτώσει και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τον έχουμε έναν προπολογισμό με 93% για επενδύσει. αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για προστιθέμενη αξία. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσουμε είναι τι να κάνουμε με τον προπολογισμό, τι θέλουμε να πετύχουμε με 1% του ΕΠ, όταν στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι περίπου το 20% του ΕΠ εκεί. Και δεδομένου των νέων προκλήσεων, των νέων πολιτικών, διεύρυνσης, το ερώτημα είναι, θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη μέθοδο και αυτό το προπολογισμό που είναι τόσο περιορισμένος ή με μια μικρή αύξηση μπορούμε και θέλουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις επιθυμίες και στις προσδοκίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Καβιθουμπάλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι στη σημερινή συζήτηση είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και διαφορετικές προτεραιότητες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει με όλες αυτές τις προτάσεις να προσπαθήσει να ε, φτιάξει μια σύνοψη, να, να δημιουργήσει ένα κοινό έδαφος, μια κοινή πρόταση. Όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση, όλοι θέλουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη που να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει κρίσεις και να ανταγωνιστεί στον, στον υπόλοιπο κόσμο. Και ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε το είπε. Ένα προπολογισμό, ένα δημοσιονομικό πλαίσιο του 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο δεν θα αρκέσει, δεν θα είναι αρκετό για να στάθουμε στο ύψο αυτών των προκλήσεων. Συμφωνώ με τον Ολλανδό συνάδελφο. Πρέπει να έχουμε αποτελεσματικό και σύγχρονο προπολογισμό. Η αποτελεσματικότητα όμως και ο εξυγχρονισμός πρέπει να υπάρχουν και στα ταμεία συνοχής και στην κοινή γεωργική πολιτική και στις πολιτικές επενδύσεων τις οποίες στηρίζουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της πρώτης πρωινή συνεδρίας και θα κάνουμε διάλειμμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κάρμεν Ηλιάνα Μιχαλτσέσκου, αντιπρόεδρο του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ γιατί με πλαισιώσατε και βοηθήσατε τα μάλλα για μια εξαιρετική καρποφόρα και φιλική συνεργασία. Δεν ξέρω κυρία Αντιπρόεδρε αν θέλετε εσείς να εξάγετε τα καταληκτικά συμπεράσματα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους ομιλητές και σε εσά, στο πρόσωπό σας, σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαιτέρως σε όσους από εσά πήρατε το λόγο και συμβάλατε ε, για τη διεξαγωγή αυτής της πολύ ε, ε, έντονης συζήτησης. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ, η πολυπληθής. Να μην ξεχνούμε ότι ο πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών, ώστε να ξαναπιστέψουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο θα είναι βιώσιμο και κοινωνικό. Το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, να στηρίζει τη συνοχή και την ε, πρόνοια, την καλή διαβίωση για περαιτέρω, ακόμα, ε, για περαιτέρω ολοκλήρωση στη συνέχεια. Έτσι ώστε και τα κράτη-μέλη αλλά και όσα φορές δεν είναι ακόμα μέλη να ε, συνεχίσουν σε αυτή την πορεία της σύγκλησης προς μια πιο ενωμένη Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω τώρα κάποια διαδικαστικά. Νομίζω ότι κάτω από το γραφείο σας βρίσκεται μία ε, σακουλίτσα με ένα μικρό δωράκι ε, της Προεδρίας. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι κάποιο μικρό κεραμικό νομίζω από ένα μέρος ε, της χώρας μας, από το Χορέζου. Ναι, μπορείτε να το βγάλετε και να το ανοίξετε, να το δείτε. Κατά τα λοιπά, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχθούμε και στο Βουκουρέστι. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ότι σας χειροκροτούν και έχουν κάθε δίκιο. Έχουν απόλυτο Επόμενο θέμα ε, της ε, ημερήσιας διάταξης είναι η 20η επέτειος του ευρώ, οι προοπτικές για το μέλλον. Να σας ανακοινώσω το πιο ευχάριστο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι τώρα. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το διάλειμμα για καφέ. Και μετά θα έχουμε το, ε, την 20η επέτειο του ευρώ. Επομένως, τεχνικές πληροφορίες. Έξα αριστερά είναι ο καφές. Κάνουμε διάλειμμα τώρα. Ευχαριστώ. Thank you very much.